Σας παρακαλώ να καθίσετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. La séance est ouverte. Η σε αρχίζει. Σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη πρώτα, έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τη διαβίβαση της υπεραστίας διατάξεως δύο αιτήσει για μεταφορές πιστώσεων 39 και 21 για ε, ποσά που θα καταβάλλονται στη Βενεζουέλα και στην Ουγκάντα. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει κατεπίον χαρακτήρας και ο κύριος Μορεσάν, γενικός εισηγητής και εγώ προσωπικά δεχθήκαμε να τα περιλάβουμε τα θέματα αυτά στη σημερινή μερίσια διάταξη. Όμως θα τεθούν σε ψηφοφορία μόνον εάν το επιτρέψει ο χρόνος διότι έχουμε ιδιαίτερα ε, επιβαρημένη, ας πούμε έτσι, ε, διαδικασία ψηφοφοριών. Στο μέλλον δε παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάζει νωρίτερα τα αιτήματα επίγοντος χαρακτήρα, ώστε να μπορέσουμε να οργανωθούμε καταλήλως. Σας ευχαριστώ για ε, την κατανόησή σας. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω στη, να σας τις αποφάσεις των συντονιστών που βρίσκονται στα πρακτικά στους φακέλους σας και αν δεν έχετε καμία ένσταση, τότε θα θεωρήσω ότι τα εγκρίνετε. Έχουμε λάβει και ανακοίνωση σχετικά με τα κοινοποίηση των πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων ε, του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου και αν δεν υπάρχει ένσταση, τα σχέδια ε, πρακτικών θεωρούνται και αυτά ότι εγκρίνονται. Μετά τα πρώτα αυτά εισαγωγικά λόγια θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία όπου αντιλαμβάνεστε όλοι και όλες την ιδιαίτερη σημασία και μιλώ για την ψηφοφορία επί της ενδιάμεσης εκθέσεως καινούρια ας πούμε ορολογία αυτή για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27 λίγα λόγια για τους ιδίους πόρους καρπός πολύμινων εργασιών ε, υπό την καθοδήγηση των ε, κ. Μπρίς και Τωμά και του κ. Λεβαντόφσκι για τους ιδίους πόρους και του κ. Ντεπρέ. Εργασίες οι οποίες έγιναν σε στενή συνεργασία με τους κοιόδης συγητές, με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και βεβαίως και με πολλές άλλες γνωμοδοτούσες επιτροπές, καθώς και με την διάσκεψη των Προέδρων Πολιτικών Ομάδων, ώστε να υπάρχουν νούμερα του Κοινοβουλίου ανά πρόγραμμα. Νέα κατάσταση αυτή και η οποία μας επιτρέπει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο Υπουργών, εάν βεβαίως τελικώ συμφωνήσει μεταξύ του το Συμβούλιο για να μπορέσει να προχωρήσει σε συζητήσεις μαζί μας. Αυτή η ενδιάμεση έκθεση, interim report, προ, προ, περιλαμβάνει και ορισμένες τροπολογίες για τον κανονισμό του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και για την διοργανική συμφωνία και θα αποτελέσει επομένω μια ιονή νομοθετική θέση του Κοινοβουλίου που θα το επιτρέψει να παρέμβει με επικοδομητικό τρόπο στην διαδικασία εγκρίσεως, consent, του μελλοντικού σχεδίου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι αριθμοί, τα αριθμητικά στοιχεία, τα νούμερα που θα ψηφιστούν θα έχουν και άμεση επιρροή στις γνωμοδοτήσεις που θα ψηφιστούν αμέσως μετά. Μετά από αίτημα της ε, ε, Επιτροπής Προϋπολογισμών. Προσκλήθηκαν όλοι οι ευρωβουλευτές να αναφερθούν στα νούμερα αυτά και να κάνουν συγκρίσεις με αυτά που θα περιλαμβάνονται στην ενδιάμεση έκθεση. Και έχουμε επομένω και τα νούμερα που θα περιλαμβάνονται στη δική μας γνωμοδότηση. Συμβαστικές τροπολογίες θα απηχούν τα νούμερα του ε, πολιτικού και έχουν μπει στις τροπολογίες. Μετά από αυτές τις διευκρινήσεις Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ορίστε κύριε Τομά. Μην ανησυχείτε, δεν είναι για να παρέμβω τις εκθέσεις. Ε, ξέχασα απλώς την ε, κάρτα ψηφοφορίας. Αυτό ήθελα να θέσω υπόψη σας. Α, και μάλιστα σε μια ιστορική ψηφοφορία. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους μου για την ε, θερμή αυτή υποδοχή των λόγων μου. Παρακαλώ βάλτε λοιπόν τώρα τις κάρτες σας στην ε, κατάλληλη σχισμή για να μπορέσουμε να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία αυτή. «25 λοιπόν ψήφισαν, μάλλον 25 κάρτες, 24 κάρτες οι 24 πρόσωπα ψήφισαν, χωρίς την κυρία Τωμά βεβαίως που δεν έχει κάρτα. Ποιο είναι 25ος. Όσοι βάλατε τις κάρτες στη σχισμή τη συσκευή. παρακαλείστε να ψηφίσετε. Ορίστε λοιπόν έγινε η ψηφοφορία, δοκιμαστική όπως είπαμε και ε, τώρα έκλεισε. Ψηφίζουμε την συμβαστική α. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 24 αποσύρεται. Συμβαστική Β υπέρ. υπέρ, κατά και αποχές. Και εγκρίνεται ε, συμβαστική Γ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Δ, D, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Amendement numéro 60, qui est pour, qui est contre. κατά αποχές και απορρίπτεται. Ε, τώρα η τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά εγκρίνεται. 66 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 16-10. Πιο σωστά 10-16. Και υπολόγισα και την ψήφο σας κύριε Τόμα. Α, βρήκατε την κάρτα. Υπέροχα. Τέλεια. Επρόκειτο για την τροπολογία 66 και πάμε στο 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 71 υπέρ κατά α, αποχές απορρίπτεται ε, 70 υπέρ κατά εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική G. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H. Ας, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78. Και έχουμε εδώ πέρα προφορική τροπολογία των εισηγητών ή συνεισηγητών υπέρ κατά εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 συγγνώμη, υπέρ κατά απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά και απορρίπτεται 88 και πάμε στο θήτα. στα ελληνικά. Ι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 συγγνώμη έχει καταπέσει και πάμε στο 132 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται Ζ δηλαδή γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κα δηλαδή γιώτα α υπέρ κατά εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική L β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπληκτή η 151 η υπαριθμό 152 επίσης 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 αποσύρεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική M δηλαδή γάμα υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 με προφορική των συνεισηγητών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 3 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά. Αποχές και εγκρίνεται. Συμβιβαστική εν, δηλαδή γιώτα δέλτα υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 174 έχει αποσυρθεί. Ε, ο, δηλαδή γιώτα ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά. Συγγνώμη, 175 που απορρίπτεται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται π, δηλαδή γιώτα σίγμα τάφ, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Nous avons terminé avec des amendements relatifs au cadre financier pluriannuel. On passe maintenant au volet ressources propres. Τώρα για τους ιδίους πόρους. Promis Q, qui est pour. Και πάμε τώρα στο Q, αποχές, εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά απορρίπτεται η ερ δηλαδή η γιώτα είδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, S γιώτα θήτα υπέρ κατά εγκρίνεται τε. κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, δηλαδή καπα υπέρ κατά εγκρίνεται Β δηλαδή καπαβίτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ κατά αποχές 208 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική W K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τρεις τροπολογίες, ε, το ίδιο αντικείμενο που είναι η προφορική τροπολογία των εισηγητών, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, εγκρίνονται. 217 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 218 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα Πανερχόμαστε στο τμήμα ε, των αιτιολογικών παράγων του πολιτού πλαισίου και έχουμε την συμβαστική ΚΔ υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ καταπίπτει αλλά όχι η 7. Όχι ψηφίζουμε το 8. Υπέρ κατά απορρίπτεται. Η γκρέκ κάπα ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το σε στα σχετικά με την ρύθμιση 237 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 237 μετά. Έχουμε κάποιες ε, τροποποιητικές που έχουν στόχο την ε, τροποποίηση της νομοθεσίας. Πρώτα απ' την ε, τροποποίηση 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροποποίηση 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροποποίηση 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 243 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροποποίηση 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροποποίηση 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 245 υπέρ κατά Α, όχι, γιατί καταπίπτει. Πάμε στο 246 που και αυτή καταπίπτει και πάμε στο 247. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρόπιση 17 με προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, α, αποχές, εγκρίνεται. «248, 249, 250 καταπίπτουν, πάμε στο 251, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, παριθμόν 20 τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 253 κατά πίπτη τροποποίηση 21 υπέρ κατά ε, υπέρ κατά 22 απορρίπτεται συγγνώμη εγκρίνεται 254 η οποία καταπίπτει και πάμε τροποποίηση 23 υπέρ κατά ε, καταπίπτει 255, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 256 καταπίπτει 257 επίσης 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 25 ε, αποσύρθηκε 259 και άλλα και αυτή καταπίπτει. Τροποποίηση 26 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 260 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ε, τροποποίηση 27 υπέρ Για το 27 ψηφίζουμε. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροποποίηση 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές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 Συμβιβαστική ΑΜΠ. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 273 τροπολογία. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογή, τροποποίηση, συγγνώμη, υπαριθμών 1. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 219 καταπίπτει. Τροποποίηση παριθμών 2 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροποποίηση 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 221 υπέρκατα, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροποποίηση 5 υπερκατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπλία 222 κατά τροποποίηση 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολόγια 3. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροποποίηση 8 υπέρ κατά εγκρίνεται Τροπολογία 24 κατά 225 επίσης 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 229 και 230 διότι είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτονται τροποποίηση 9 υπέρ κατά εγκρίνεται συνδεστική ΑΣΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροποποίηση 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική αντέ. υπέρ. Κατά. Εγγύηση. Ε, τροποποίηση 12 εγκρίνεται. Αύκο. Τροποποίηση 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η επόμενη, ε, η 13 απορρίπτωτη και τώρα έχουμε αυτές τις προτάσεις για μια διοργανική συμφωνία και έχουμε την τροποποίηση 46 υπέρ, κατά, ε, αποχές, εγκρίνεται. Σε τροποποίηση 47 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Καταπίπτει η τροπολογία 274 ψηφίζουν την 275 υπέρ κατά απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει τροπολογία 276 τροποποιεί 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 277 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται τροποποίηση 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροποποίηση 53 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 278 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροποποίηση 54 έχει αποσυρθεί 55 υπέρ κατά εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 279 κατά πίπτη 280 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 281 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 282 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 283 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 284 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 285 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροποποίηση 53, 57, συγγνώμη, 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 286 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροποποίηση 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 287 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 288 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροποποίηση 60 έχει αποσυρθεί. Πάμε στο 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροποποίηση 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στα παραρτήματα ε, και καλύπτονται από την συμβαστική ΑΕ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Και επομένως τώρα θα πάμε απευθείας στο συμπέρασμα. Γιατί όσον αφορά τα παραρτήματα έχουμε τις παραδεκτές τροπολογίες οι οποίες καλύπτονται από την συμβαστική γιατί πρόκειται για κάποιες προτάσεις ε, τις που είτε καλύπτονται είτε είναι απαράδεκτες. Οπότε πάμε τώρα να δούμε το σύνολο αυτής της προσωρινής εκθέσεως ακριβώς όπως έχει τροποποιηθεί. Θα γίνει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ονομαστικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 25-5. Χωρίς αποχές. Τα χειροκροτήματα εκφράζουν τα θερμά συγχαρητήρια για τους τέσσερις συνεισηγητές αλλά και τους σκιώδεις εισηγητές, οι συνεισηγητές. Να πώς βλέπουμε το ότι τώρα είναι σαφής η εντολή και τώρα έχουμε να κάνουμε το Συμβούλιο. Une étape importante et que nous avons pris les dispositions pour que la négociation s'engage sur des γιατί θα πρέπει τώρα να πάμε σε διαπραγματεύσεις ε, με ξεκάθαρη εντολή. Θα πρέπει να δούμε το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά αναπρόγραμμα. Τώρα θα πρέπει να κρίνουμε την ετησία έκθεση της Έντερ Γκαρτιαθάβαλ όσον αφορά τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τροπολογία 1 με προφορική τροπολογία. Παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 λέει ο πρόεδρος, αλλά εννοεί 9 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ, 14 κατά. Και μία αποχή. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αποσύρεται ή μάλλον έχει αποσυρθεί η 14 συμβαστική σ γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εδώ θα χρειαστεί επαλήθευση συμβαστική 20 με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος η τροπολογία 20 συγγνώμη η τροπολογία 20 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με ψήφους 18 κατά 11 υπέρ Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ήθελα να επαναληφθεί. 21 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά δεν είναι σαφές για το 23, για 23 λοιπόν. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Τέλος. Ψήφι 19 υπέρ, 11 κατά. Ήταν λοιπόν 23. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται «29 υπέρ» κατά αποχές εγκρίνεται «30 υπέρ» κατά θα επαληθεύσουμε εδώ λοιπόν η 30. Τέλος της ψηφοφορίας. Ψήφι 13 υπέρ, 16 κατά. Τροπολογία υπάρχουν 30 υπέρ. Με συγχωρείτε, 31, 31. 31 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία η οποία αρχίζει. Τέλος, εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ, 4 κατά και συγχαίρω την κυρία Γαρδιά Θαμπάλ. Τώρα θα συνεχίσουμε με την έκθεση του κ. Γκέρενς. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές όμως το αποτέλεσμα. Θα, αρχίσουμε, θα κάνουμε λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται ψήφι 23 υπέρ, 6 κατά. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια, μην διστάζετε. Τροπολογίες 5 και 6, ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές, αποσύρονται λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 5 και 6. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, ας, επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψήφος επαληθεύσεως. Πέρας. Μάλιστα και μαζική ψήφος υπέρ. Παρακαλώ σηκώνετε καλά τα χέρια. Τροπολογίες 7 και 8 είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τώρα, για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει, τέλος, εγκρίνεται ψήφι 24 υπέρ, 6 κατά. Και συγχαρητήρια κύριε Γκέρενς. Έχουμε τώρα τις γνωμοδοτήσεις για τα διάφορα δημοσιονομικά προγράμματα και θα κάνουμε μια πρόταση. Υπάρχουν πλήρωνες συμβαστικές τροπολογίες για την ενδιάμεση έκθεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τους στόχους του κλίματος με την εξής διατύπωση η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον στόχο προστασίας του κλίματος θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στο 25% των δαπανών του ΠΔΠ 2021 έως 27 και 30% το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από το 2027. Άρα υπάρχουν δύο επίπεδα. Ένας συνολικός στόχος επταετίας με τουλάχιστον 25% και ένας στόχος ετήσιος για να φτάσει ο στόχος το δυνατόν συντομότερο στο 30% και το αργότερο πάντως μέχρι το 2027. Θα ε, ψηφίσουμε διάφορες τροπολογίες που αναφέρονται σε ένα συνολικό στόχο του 30%, κάτι το οποίο βέβαια έρχεται σε αντίφαση με την ενδιάμεση έκθεση που μόλις ψηφίσαμε προηγουμένως. οι εισηγητές και συντάκτες τροπολογιών έχουν περιλάβει και προφορική τροπολογία για να περιληφθεί η συμφωνημένη διατύπωση στην ενδιάμεση έκθεση. Και τους ευχαριστώ. Ωστόσο, οι τροπολογίες αυτές έχουν ένα καταρχήν αντιφατικό χαρακτήρα, γιατί έχουμε ορισμένες τροπολογίες για το πρόγραμμα LIFE, για αξίες, για την τροπολογία 18, για την παγκοσμιοποίηση. Αυτές οι τροπολογίες έχουν όλες υποβληθεί από την κυρία Γιάντεν Μάκη, η οποία δυστυχώς σήμερα κολλείεται. Αν δεν έχετε κάποια ένσταση, κυρίες και κύριοι, και για να υπάρξει μια συνεκτικότητα στις ε, τροπολογίες αυτές που θα ψηφιστούν τα επόμενα λεπτά, θα προτείνω να ληφθεί υπόψη μια προφορική τροπολογία που επιγράφεται κλίμα με το εξή κείμενο. ένα συνολικό στόχο του 25% των δαπανών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την υποστήριξη κλιματικών στόχων στα πλαίσια του ΠΔΠ 21-27 και ένας ετήσιος στόχος του 30% τον συντομότερο και πάντως το αργότερο μέχρι το 2027. Συμφωνείτε με αυτή την ε, πρόταση, τη διαδικαστική πρόταση. Έχει καλώς. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ε, δηλώνω ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την συμφωνία σας. Τώρα, για, το, για την πρώτη ψηφοφορία, για τη συνεργασία στα τελωνία. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, με προφορική τροπολογία αυτή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. για τι αιτιολογικές σκέψεις. Ε, τροπολογία πέντε υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι αποσύ... απορρίπτεται, συγγνώμη, αλλά ας επαληθεύσουμε καλύτερα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται όντω. Ε, τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψήφος. Πέρας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ και 2 κατά και συγχαίρω τον εισηγητή. Τώρα το πρόγραμμα φυσκάλης. Τροπολογία 8 υπέρ. Για το κείμενο φυσκάλης. 8 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 να με συγχωρείτε για το θόρυβο. Θα φροντίσω να μην επαναληφθεί. ε, ε υπέρ κατά αποχές. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 συμβατεί με την 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται.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 5 υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται ότι απορρίπτεται αλλά ας επαληθεύσουμε τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται όντως με ψήφους 18 κατά 11 υπέρ Προπολογία 14 υπέρ. 13 λέτε. Μόλις ψηφίσαμε, μόλις απορρίψαμε την 5. Η 13 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται για το σύνολο του κειμένου. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. 24 ψήφοι υπέρ, 5 κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Συγγετρία. Για την κυρία Γιατενμάκη τώρα, για το πρόγραμμα Life Τροπολογία 23. Υπέρ, κατά, αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψήφος. Ψηφίσατε. Τέλος. Απερίφθη. Ψήφι 16 κατά, 13 υπέρ. Τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 το μπορούν να ψηφιστούν όλες μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Α, επιθυμείτε να γίνει επαλήθευση. Από την 2 έως την 8 αρχίζει. Εγκρίνονται 18 ψήφοι υπέρ 12 κατά. Τροπολογία 24. Α, καταπίπτουν αυτοί. Ωραία, προχωρούμε στην 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Και 1. Επανερχόμαστε στην τροπολογία για το κλίμα, με την επιγραφή κλίμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για τις αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ, κατά Ας επαληθεύσουμε την 14. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Ψήφι 20 υπέρ 10 κατά. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 έχει αποσυρθεί. 10. Με συγχωρείτε. Α, πηγαίνουμε στην 19. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Άρα, προχωρούμε αμέσως. Α, προχωρούμε στην τελική ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος, με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Τέλο εγκρίνονται, με 26 ψήφου υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Γιάτεν Μάκη. Έκθεση Λαμασούρ για το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμήνη. 44 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σαράντα 5 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 47 καταπίπτει. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 49 καταπίπτει 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 ε, 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 52 ε, καταπίπτει 3 Ναι, ναι, συμβατή. Υπέρ λοιπόν τη 52, λέει ο τώρα, 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 ε, αυτή εκπίπτει μια στιγμή όχι, όχι 55 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εδώ θα επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 6. Τέλος της ψήφου. Ψήφι 18 υπέρ, 10 κατά και μία άποχη. Η 6 εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 62, 63 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψήφο. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψήφι 17 κατά 12 υπέρ. 68 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εδώ θα επαληθέσουμε διότι δυστυχώ δεν σηκώνονται καλά όλα τα χέρια 71 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται ψήφι 17 υπέρ και 12 κατά 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ. Παρακαλώ, σηκώστε καλά τα χέρια. Ή ε, τώρα ή μετά θα τα σηκώσετε. 8 λοιπόν υπέρ. Κατά. Δεν σηκώθηκαν όλα τα χέρια. Άρα δεν θα αποφύγουμε την επαλήθευση για την ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για την 8. Πέρας εγκρίνεται με ψήφους 17 υπέρ και 11 κατά. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά μεγάλη χάρη θα μου κάνετε αν σηκώνετε πραγματικά καλά τα χέρια. Όπως θέλετε υπέρ ή κατά. Για την 9 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10. Θέλετε τσεκ για την 9. Καλώς. Αρχίζει η ψηφοφορία επαλυτεύσεως. 9, ε. Πέρας. Εγκρίνεται με ψήφους 16 υπέρ, 11 κατά. Προπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά εγκρίνεται για τις αιτιολογικές σκέψεις 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο με υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με συγχωρείτε 23 υπέρ. Επαναλαμβάνω. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. με ναι, κάποια έκπληξη στη φωνή. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά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 δεν είναι απόλυτα σαφές η ηλεκτρονική παρήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται με ψήφους 18 υπέρ, 9 κατά. Ήταν λοιπόν η 33. 34 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 και 40 με προφορική τροπολογία του εισηγητού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εγκρίνονται μάλλον. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά εγκρίνεται. Για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει ψηφίσατε άπαντες πέρας εγκρίνεται με ψήφους 22 υπέρ 5 κατά συγχαρητήρια κύριε Λαμασούρ. Alors, on en vient au contrôle. Πάμε τώρα στον συνοριακό έλεγχο. Χολμάιερ. 30, 45 και 16 μαζί υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9, 10, 11, 12 και 13 ε, όλες μαζί υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία υπαριθμών 40 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, δεν σηκώσατε όλοι τα χέρια. Επομένως πάμε για ηλεκτρονική ψηφοφορία και ψηφίζουμε. Δεκαέξι, δέκα, μία αποχή εγκρίνεται. 41 ένα, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίβεται. 42 δύο, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται 43 δεν έχω ψήφο 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 έλεγχος για το 46 ψηφίζουμε πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 15-12. Καλά τα λέγατε. Ε, πρόκειτο για την 46 47. Πού εγκρίνεται 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ σηκώστε ευκρινώς το χέρι σας. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά απορρίπτεται 20 υπέρ κατά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 η επόμενη. 28. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σόφρα το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 23-2. Συγχαρητήρια Μόνικα. Και τώρα. Έχουμε την ε, έκθεση Κίρτσου. Sur les, aux, aux Στον αφορά το, τον εξοπλισμό ελέγχου για τα τελωνία. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6, 7, 8, 9 και 10 όπως και το 12 και το 1 όλα αυτά από κοινού υπέρ υπέρ κατά αποχές qu'ils sont εγκρίνεται 22 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Και pour. Και Περ κατά αποχές και εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. 14 αποσύρεται. 22. Υπέρ. Όχι, συγγνώμη, λοιπόν, οι δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά ας κάνουμε επαλήθευση με ονομαστική ψηφοφορία όχι συγγνώμη λάθος με ηλεκτρονική ψηφορία διορθώνει ο πρόεδρος ψήφισαν όλοι πέρα ψηφορίας Α, απορρίπτεται 10 18 υπάρχει μόνο 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές το, σύνολο τώρα του κειμένου όπως ε, τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε Σκοτάει κλού Πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται 25-2 και μία αποχή και τώρα έχουμε την επομένη έκθεση είναι η έκθεση Μορέν. Όσο αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 39. Υπέρ κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Το 42 έχει αποσυρθεί. Το 43 συμβατό. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 9. Πρώτο τμήμα. Καλύπτεται από την συμβαστική 1. Οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά. Βλέπω ότι δεν σηκώνετε ευκρινώς τα χέρια σας γιατί μάλλον κουραστήκατε. Ξαναρωτώ, ποιοι είναι υπέρ του δευτέρου τμήματος του 9, υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται 49, υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται 47, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 48, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 50. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51, υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ας κάνουμε επαλήθευση για το 52 ηλεκτρονικά ψηφίζουμε πέρας 8-19 απορρίπτεται 53 προφορική τροπολογία υπέρ κατά δεν έχετε σηκώσει όλοι τα χέρια άρα έχουμε για το 53 επαλήθευση ηλεκτρονικά ψηφίζουμε ψηφίζουμε πέρας και απορρίπτεται 12-15 13 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 54 Κυρία Τωμά θέλετε το λόγο όχι λέει κυρία Τωμά Non, vous ne souhaitez pas vous exprimer. Alors... Εφού θέλετε να μιλήσετε, μιλούμε για το 54. Καταπίπτει όπως και το διακόπτει ο πρόεδρος. Α, ah. bon. Alors, comme, comme le 53 est... Α, μάλιστα, δίκιο έχετε το 54 πέρασε από ηλεκτρονική ψηφορία. Οπότε και το 53 θα πρέπει να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Merci. Ευχαριστώ, με διορθώσατε. Πέρας της ψηφορία για το 53.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 repoussé par 15 voix contre 14. Και απορρίπτεται 14-15. 14. 14 14 με προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Il a voté pour. Ils ont une vieille liste de vote qui avant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 για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Ψηφίζουμε. Oui. Scrutin est clos. Approbation par 22 voix contre 5. Και εγκρινεται 25. Le 59 qui est compatible avec le 14, qui est pour. Παρακάτω, το 59 είναι συμβατό με το 14, υπερκατά αποχές και απορρίπτεται το 59. Και πάμε στο 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και Και contre. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 66, υπέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 έχει αποσυρθεί. 70 υπέρ κατά απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στις ιδεολογικές παραγράφους. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για το 18. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Σκοτάει κλου. Πέρα Και απορρίπτεται 10, 17, 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 23 και 24 διότι είναι ταυτόσιμες. 23 και 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 25 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ψηφίζουμε. Και εγκρίνεται 15-13. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28. Και 29. Είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά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 εγκρίνεται 38 υπέρ κατά εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε μας και ψηφοφορία ψηφίζουμε πέρα ψηφοφορίας 24-3 εγκρίνεται. Υπάρχει και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Γκλόνεκ. Έκθεση Σολέ. Για δικαιώματα και αξίζει η τροπολογία. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 7 θα καταπέσει γιατί καλύπτει. 28 υπέρ κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για επαλήθευση. Για το 28. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Και απορρίπτεται 13-15. Το 8 απορρίπτεται, πάμε στο 13. 30 εννοεί ο πρόεδρος. Pardon, παρδόν, pardon. Αχ, συμπαθάτε με λέει. Ευτυχώ που έχω και εσά. 30, 30. Και όχι 13. Υπέρκατα Αποχέ. Να κάνουμε υπαλήθευση. Για το 30. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 11-17 31 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 31 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 16-12 ή 12-16 το 9 αποσύρεται Παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε μαζί. 29, 21, 24, 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτονται 11-17. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά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 Εψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται 8, 10, 9. και το 46 και το 47 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές παράγραφοι 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεκαεννέα. Υπέρ. Για το κλίμα, ε, αναφέραμε την προσωπική τροπολογία. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. υπέρ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με την ψηφοφορία ψηφίζουμε. Πέρασε. Και εγκρίνεται 24-4 χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σολέ. Γκοντζάλες Πόνς. Euh, Πρόγραμμα για την δικαιοσύνη. Τροπολογία 5 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για τις αιτιολογικές σκέψεις 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή στο σύνολο του κειμένου ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει Πέρας. Εγκρίνεται. Ψήφι 24 υπέρ, 3 κατά. Και συγχαρητήρια κύριε Κουντζάδε Πόνς. Έκθεση Μανουέλ Δος Σάντος για το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Τροπολόγια 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές ασαφές το αποτέλεσμα επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει πέρας απορρίπτεται ψήφι 19 κατά 9 υπέρ 23 υπέρ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 εγκρίνεται. Α, επαλήθευση. Επαλήθευση για τη 15 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απεριφθεί. 18 ψήφι. κατά, 10 υπέρ. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 με προφορική τροπολογία για το κλίμα υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρόκειται για εκείνη την ε, τροπολογία συνοχής, για την εξασφάλιση συνεκτικότητας δηλαδή. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Ναι, ναι, διορθώστε τις ψηφοφορίες, λέει ο πρόεδρος. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψήφι 23 υπέρ, 5 κατά. Το σύνολο τώρα. Επί του συνόλου του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει η ψηφοφορία, ονομαστικά, ονομαστική ψηφοφορία. Προλαβαίνω να πιω μια κουλιά. λέει ο πρόεδρος. Πέρα στις ε, ψηφοφορίες εγκρίνεται με ψήφους 24 υπέρ, 3 κατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Ντός Σάντος. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει, εισερχόμενος. Πρόεδρος. Φαίνεται πως δεν θέλησε να επηρεάσει την ψήφο. Έκθεση της κυρίας Βάιντερε για το Ταμείο Αλληλεγγύης για την Λετωνία. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψήφο. Αρχίζει. Ψηφίσατε άπαντες. Όχι ακόμη. Πέρας πάντως. Ψήφι 27 υπέρ, ένας κατά. Μία ψήφος δηλαδή κατά. ça c'est bien, oui. Bien, nous avons maintenant deux... Έχουμε τώρα δύο εκθέσεις. Του Πάουλ Ρούμπικ, πρώτη έκθεση για το ψηφιακό ε, πρόγραμμα περίοδου 2021-2027. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. 17. Πέρας εγκρίνεται με ψήφους 15 υπέρ, 14 κατά. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι θα χρειαστεί ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. ίδια πλειοψηφία 15 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι απόλυτα σαφές. 21 λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει. Πέρας. Πάλι 15-14. Έχουμε τώρα τις 4, 21, 22, 23, με συγχωρείτε, όχι, μέχρι τις 27, 27, που μπορούν να ψηφιστούν δια μιας. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η 7 τώρα, τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. 28. Ψηφίσατε άπαντες. Πέρασε. Ψήφι 16 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 και 30 με προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται.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 σχεδόν, λέει ο πρόεδρος, πέρας, ψήφι 27 υπέρ, 2 κατά και συγχαρητήρια στον Πάουλ Ρίμπικ. Τώρα, πάλι του ιδίου, έκθεση περί ανταγωνιστικότητας για το πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς. Τροπολογία 16. Υπέρ κατά αποχές με ονομαστική ψηφοφορία λέει ο πρόεδρος ενώ η ηλεκτρονική επαλήθευση μάλλον πέρας απορρίπτεται ψήφι 10 υπέρ 19 κατά τροπολογίες 1, 2 και 3 όλες μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α μάλλον. Στο παράρτημα τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται για τις ιδεολογικές σκέψεις τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ. Κατά αποχές ασαφές το αποτέλεσμα επαλήθευση 12 για την 12 αρχίζει πέρας απορρίπτεται με ψήφους 17 κατά 13 υπέρ τροπολογία 13 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Θα χρειαστεί παλήθευση, ηλεκτρονική παλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Της 13. Πέρας. Απορρίπτεται με ψήφους 18 κατά, 12 υπέρ. Τροπολογία 14, καθώς και 15 μπορούν να ψηφιστούν μαζί με μια προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται στο σύνολο το, το κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία η οποία αρχίζει πέρας εγκρίνεται με ψήφους 27 υπέρ κατά και συγχαρητήρια. Έκθεση που ίσως να μην χρειαστεί να την ψηφίσετε και ο Άσουερς είναι, κολλείεται δυστυχώς σήμερα το απόγευμα και παρακαλεί να προσπαθήσω να τα πω εγώ θα, θα, θα χειριστούμε όλες τις μεταφορές πιστώσεων όπως προβλέπει ο κανονισμός. Έχετε προ ημέρων λάβει όλη τη σχετική τεκμηρίωση για τις συγκεκριμένε αυτές πιστώσεις, μεταφορές πιστώσεων. Πρόκειται για τον προϋπολογισμό 2018 και μεταφορές πιστώσεων σε άλλα τμήματα. Και πρώτα για το ελεγκτικό συνέδριο, τέσσερις μεταφορές ε, πιστώσεων, τρεις εξ αυτών έχουν περιορισμένη σημασία. Πρόκειται για το κονδύλιο της ασφαλείας 27.000 ευρώ, μετακομίσεων για συντήρηση, για εργασίες συντηρήσεως 30.000 ευρώ και κονδύλιο για την τεκμηρίωση και βιβλιοθήκες 10.000 ευρώ. Τέταρτη μεταφορά πιστώσεων για δύο κονδύλια για ηλεκτρονική τεχνολογία 700.000 ευρώ. Έχουμε επίσης μεταφορές πιστώσεων για την Επιτροπή Περιφερειών και για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Πρώτα για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 983.000 ευρώ σε πλοίωνα κονδύλια για την κτήση ακινήτων, μισθώματα, τεχνικό εξοπλισμό κλπ. Η NF6 και η NF7 της Επιτροπής της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για αγορά εξοπλισμού κλπ. 763.000 ευρώ και δύο ακόμη μεταφορές πιστώσεων της Επιτροπής Περιφερειών για αποστολές με ένα ποσό και επίσης για μελέτες που ανατίθεται στο εξωτερικό 149.003 ευρώ. σκιώδεις επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Εάν όχι, εάν δεν ζητούνται διευκρινήσεις ενδεχομένως που θα μπορούσε να μας δώσει η κυρία Σάντσες Λόπες, επικεφαλής ε, του Τμήματος Λογαριασμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ο κύριος Γιάκοψεν ή ο κύριος Ρέντες για την Επιτροπή Περιφερειών, θα θεωρήσω ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις εκ μέρους σας και επομένως θεωρώ ότι εγκρίνονται οι μεταφορές πιστώσεων από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου. Ορίστε παρακαλώ. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι δεν θα ψηφιστούν. Είμαστε όμως κατά των πιστώσεων αυτών, κατά των μεταφορών πιστώσεων. Ο Πρόεδρος, σημειώνω την παρατήρησή σας, ωστόσο δεν προβάλλεται ένσταση και θεωρώ λοιπόν ότι όντως εγκρίνεται η, εγκρίνει μάλλον η Επιτροπή Προϋπολογισμών, σημειώνω βεβαίως την θέση σας. Ο Γενικός Εισηγητής επιθυμεί να τοποθετηθεί τώρα για τον προϋπολογισμό του 2018 και να μας παρουσιάσει δύο μεταφορές πιστώσεων που έχουν τεθεί υπόψη μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από την διαβίβαση της ημερησίας διατάξεως, του σχεδίου ημερησίας διατάξεως. Νομίζω ότι έχουμε επαρκή χρόνο και θα μπορέσουμε έτσι να ανταποκριθούμε στην επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Μουρεσάν. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Πράγματι υπήρξαν δύο αποφάσεις τη Επιτροπής για τέτοιες αιτήσει μεταφοράς, 29 και 31 συγκεκριμένα. Και σε τι αφορούν. Σε 42 εκατομμύρια ευρώ που θα, για να διατεθούν για την Βενεζουέλα και την Ουγγάντα. 27 εκατομμύρια για την Ουγγάντα λόγω των ε, προβλημάτων ε, σε επίπεδο επισυντηστικό και υγειονομικό. Και φαντάζομαι γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ θα ε, κατευθύνονται προ την ΟΚΑΤ. Το πρώτο λοιπόν προσωπικό για την Βενεζουέλα. Από που θα προέλθουν τώρα αυτά τα 42 εκατομμύρια ευρώ. 31 εκατομμύρια από το Emergency ε, Aid Reserve, 7 εκατομμύρια από μεταφορές από το EDCI ε, και 4 εκατομμύρια από τον ε, μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Νομίζω πως θα πρέπει να εγκρίνουμε αυτές τις μεταφορές γιατί σε κάθε περίπτωση χρειάζονται, είναι αναγκαία αυτά τα κονδύλια αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να παρακαλέσω την Επιτροπή στο μέλλον να μας ε, υποβάλει τα εν λόγω αιτήματα μεταφορών νωρίτερα. Ε, υπήρξε λοιπόν η υποβολή πριν από 10 ημέρες, δηλαδή ε, όχι την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή πριν, αλλά επειδή είχαμε την πράσινη εβδομάδα ε, διάμεσα, δεν ήταν εύκολο να προχωρήσουμε. Ε, οπότε, ε, αν υπάρξουν τέτοιε αιτήσει για αμφιλεγόμενα ζητήματα στο μέλλον, θα έχουμε προβλήματα. Ε, το συγκεκριμένο προβλήμα δεν ήταν αμφιλεγόμενο, οπότε δεν υπήρξε θέμα. Αλλά εάν υπάρξει ένα τέτοιο αίτημα στο μέλλον και υπάρξουν ε, διαφορετικέ απόψει, θα έχουμε προβλήματα. Οπότε, πρόεδρε, εξήγησα περί τίνο επρόκειται. Η δική μου πρόταση είναι να υπερψηφίσουμε αυτέ τι αιτήσει τη Επιτροπή και βέβαια θα ήθελα να ακούσω και του συναδέλφου. Σα ευχαριστώ κύριε Γενική Εισηγητά. Νομίζω ότι σημειώνει την ε, παράκλησή σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλωστε την είχα επαναλάβει και εγώ στην αρχή της σα, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να κάνει έγκαιρα τις αιτήσει μεταφορών πιστώσεων, ώστε να ε, σεβόμαστε και την σοβαρότητα, που δεν έπασχε εν προκειμένου, διότι τελικώς δέχεται με την γνωμοδότησή του και ο Γενικός Συγητής. Θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα με ονομαστική, μάλλον με ηλεκτρονική ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρο. Αρχίζει η ψήφος. Ψηφίσατε άπαντες. Περιμένω λίγο ακόμη. Ίσως κάποιος βγήκε έξω αφήνοντας την κάρτα του στη σχισμή. Ε, πάντως τώρα έληξε η ψηφοφορία. Έχω λοιπόν 20 ψήφους, 18 υπέρ και 2 κατά. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εγκρίνει τις σχετικές μεταφορές πιστώσεων. Η Νικόλ Μεγιέρ δεν έχει να μας ανακοινώσει. Α, συγγνώμη, η κυρία Χόλμαϊερ, ε, δεν είχε να ανακοινώσει τίποτε σχετικά με την ε, πολιτική ε, κτίριων. Δεν έχουμε άλλη ψηφοφορία, δεν έχουμε οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με την κτηριακή πολιτική. Θα δώσω πάλι το λόγο στον κύριο Μουρεσάν για να κάνει την παρουσίαση του διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 6 για το οικονομικό έτος 2018. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. το σχέδιο λοιπόν διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 6 για το οποίο σας υπέβαλα την ε, σχετική έκθεση ε, αφορά στο εξή. Ε, συνήθως αυτή την περίοδο του έτους, όπως δηλαδή συνέβη και πέρυσι και πρόπερσι, η Επιτροπή πρέπει να προετοιμαστεί και να κάνει ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δώρο προς τα κράτη-μέλη προκειμένου να αυξηθεί η απορρόφηση των κοντιλών που τους έχουν διατεθεί. Αυτό έγινε πέρυσι και πρόπερσι. Ε, φέτος τα πράγματα ωστόσο είναι πολύ καλύτερα, δηλαδή η ολοποίηση έχει προχωρήσει καλύτερα, τα project τρέχουν με πλήρη ε, ρυθμού ταχύτητα, οπότε τα αποτελέσματα που βλέπουμε φέτο είναι καλύτερα σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι. Άρα λοιπόν αυτό το ε, DAP προ... Ε, μία ε, μείωση ε, κατά 48,6 εκατομμυρίων των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 44,7 των πιστώσεων πληρωμών. Κατά τα λοιπά, έχουμε να κάνουμε με τις δαπάνες. Ό,τι αφορά την πλευρά των εσόδων, υπάρχει μία επανεξισορρόπηση των όσων προτείνονται στο προπολογισμό της Ένωσης. Μιλάμε δηλαδή για μία τεχνική και αυτόματη διαδικασία, η οποία σε τι αφορά στο ότι υπάρχει μία μείωση των καθαρών δασμών που σε ε, τα κράτη-μέλη ε, της τάξης των 2,6 δις ευρώ. Και υπάρχει και επίσης ε, μία αναπροσαρμογή στο επίπεδο των 90 εκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά τη βάση του ΦΠΑ. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, εάν τα έσοδα από τους ίδιους πόρους είναι χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονταν, αυτόματα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, προβούν στην ε, συμπλήρωση, αν θέλετε, με βάση την δική τους εθνική συνεισφορά ε, και κατά συνέπεια αυτή είναι η αλλαγή. και με βάση το όσο προβλέπονται, τα όσα προβλέπονται από τα κράτη, για τα κράτη-μέλη, με βάση δηλαδή τους ιδίους πόλους που θα πρέπει ε, να ε, ε, υποβάλουν. και βέβαια υπάρχει και η περίπτωση των 8 εβδομάδων τώρα σε ό,τι αφορά τη συνδιαλλαγή με τα εθνικά κοινοβούλια. Από εκεί και μόνο μετά θα γίνει μια ψηφοφορία. Δηλαδή αναμένω την ψηφοφορία εδώ στο κοινοβούλιο μα το Δεκέμβριο. Αλλά από την δική μου πλευρά, Πρόεδρε, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για τεχνικό ζήτημα, το έχουμε συζητήσει ή το είχαμε συζητήσει κατά το τελευταίο τριμερή διάλογο με το ε, Συμβούλιο και με την Επιτροπή, οπότε δεν προβλέπω να προκύψει κάποιο πρόβλημα και όπως είπα θα, το, θα ψηφιστεί αυτό το ζήτημα τον Δεκέμβριο. Ευχαριστώ. Merci, le Ευχαριστούμε κύριε Γενική Εισηγητά. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, όχι. Επομένως, το ραντεβού μας για αυτό ανανεώνεται για τις 19 ενδεκάτου, ούτως ώστε να γίνει μέχρι τότε η κατάθεση των τοπολογιών. Όριο είναι 6 ώρα το απόγευμα και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 21 Ενδεκάτου. Ούτως ώστε το κείμενο να κατέβει στην Ολομέλεια στην ε, δεύτερη σύνοδο του Νοεμβρίου. Mobilisation. Ε, τώρα το θέμα αυτό το επόμενο αφορά την κινητοποίηση, δηλαδή ενεργοποίηση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφυγών στην Παγκοσμιοποίηση και η συγκεκριμένη είναι η κυρία Καρδία Θάμπολ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα θα σα τα πω γιατί βλέπω ότι όλο ένα και λιγότεροι είναι οι παρόντε ε, εδώ γιατί είχαμε τόσε τόσε ψηφοφορίε. Πότε έχουμε εδώ πέρα την ε, ε, λόγο αίτηση στο Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και είναι η δεύτερη φορά που η περιφέρεια τη Αττική και για τον ίδιο κλάδο των εκδοτών ζητεί την ενεργοποίηση του Ταμείου. Μιλούμε για κάποιες ε, απολύσεις 550 από τρεις διαφορετικές ε, εταιρείες και θα έχουμε κάποια ενίσχυση που θα είναι της ε, τάξης του 60% του συνολικού δηλαδή 2,3 εκατομμύρια. Οπότε βλέπετε ότι οι πράξεις που προβλέπονται είναι σημαντικές και αυτά όλα αποφασίστηκαν σε συντονισμό με τους φορείς των δημοσιογράφων αλλά και το Υπουργείο Απασχόλησης. Δόθηκε το πράσινο φως, επομένως δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Merci. Ο Πρόεδρος, εμείς σας ευχαριστούμε για τα όσα μας είπατε τα που ήταν τόσο ενθαρρυντικά. Ζητεί κανείς το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. 6 11. Αύριο δηλαδή ε, το μεσημέρι είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες και πρώτα να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 21 και ε, θα κατέβει το θέμα στην Ολομέλης κατά την δεύτερη σύνοδο του Νοεμβρίου. Και τώρα. Γιάννης Γκάιερ, στρέφουμε προς ε, εσάς σχετικά με τον έλεγχο των αποκεντρωμένων οργανισμών. Είναι δική σας γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην πλούσια γερμανική γλώσσα υπάρχει αυτό το ρητό ότι ε, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε και σε μια άδεια αίθουσα και θα, θα δω πώς λειτουργεί στην πράξη αυτό το ρητό. Ε, αναφερόμενο σε αυτό το ζήτημα των αποτιτρωμένων οργανισμών, ε, το οποίο σίγουρα αποτελεί ένα πολύ γοητευτικό ζήτημα. Ο συνάδελφος Μπον Σλόπφλιν είχε αναλάβει ε, ή έχει αναλάβει να συντάξει με σχετική έκθεση και εγώ, επειδή είμαι αρμόδιο για αυτά τα ζητήματα από την πλευρά της Επιτροπής Επιτροπή Προεπολογισμών αποφάσισα ότι κάτι τέτοιο, μια τέτοια δηλαδή γνωμοδότηση θα πρέπει να συνταχθεί χωρί την δική μας άποψη, χωρί τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προεπολογισμών. Άρα λοιπόν ε, θα ήθελα καταρχήν ε, να καλέσω όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται, ε, για αυτό το θέμα να κάνουν τα δικά τους σχόλια γιατί εγώ έχω συντάξει μια πολύ σύντομη γνωμοδότηση ε, επειδή με περιορίζει το καταστατικό του Κοινοβουλίου στο να περιοριστώ στα βασικότερα ζητήματα. Καταρχήν, ε, αναφέρομαι λοιπόν σε αυτή τη γνωμοδότηση στο ζήτημα της χρηματοδότησης των τελών, ένα ζήτημα δηλαδή που έχει προκύψει επανειλημμένα και ε, αναφέρω ότι πρόκειται στο διάμεσο διάστημα πλέον για ένα δισεκατομμύριο ευρώ ε, το οποίο θα μπορούσε δηλαδή να ειστρέψει στον κορβανά αυτών των αποκυρωμένων οργανισμών μέσω των τελών, εάν για παράδειγμα υπάρχει χρέωση τελών απέναντι για παράδειγμα στον κλάνο. σε, δηλαδή σε αυτούς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς ε, αυτού του είδους, ε, αυτού του κλάδου. τώρα, ένα ακόμα ζήτημα που μας έχει από απασχολήσει επανειλημμένα είναι βέβαια αυτό της έδρας των οργανισμών το οποίο αφορά και ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη. Ε, στο παρελθόν υπήρξαν κάποια ζητήματα σε σχέση με αυτό, δηλαδή ότι ε, κάποιοι οργανισμοί τελικά είχαν περισσότερες ε, από μία έδρες, ενώ υπήρξαν και υπηρεσίες των οποίων η έδρα βρίσκονταν σε πολύ απομακρυσμένα σημεία ή βρίσκεται ακόμα σε πολύ απομακρυσμένα σημεία και βέβαια με αυτό το θέμα σχετίζεται και ένα ακόμα πρόβλημα. Εάν δηλαδή δεν υπάρχει για παράδειγμα ένα διεθνές σχολείο κοντά στην έδρα ενός αποκεντρωμένου οργανισμού, ε, τότε ε, είναι δύσκολο για παράδειγμα να εξευρεθεί και το αρμόδιο ε, προσωπικό με την κατάλληλη προγνωμοσύνη και εμπειρία γιατί ακριβώς δεν έχουν που να στείλουν τα παιδιά τους για το καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε εδώ είναι καλέσουμε την Επιτροπή σε σχέση με εκείνους τους οργανισμούς οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν διπλή έδρα ε, ε, να κάνει μια αξιολόγηση ως προς το κατά πόσο κάτι τέτοιο εξακολουθεί να είναι απαραίτητο. Ε, κάτι ακόμα που αναφέρω στη δική μου γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά το προσωπικό είναι ο συντελεστής της τροποποίησης. δηλαδή σε ό,τι αφορά τα νέα κράτη-μέλη γνωρίζετε ότι εφαρμόζουμε ένα ε, μισθολογικό συντελεστή ε, σε ό,τι αφορά το προσωπικό του, το οποίο βέβαια συντελεστής ε, του εποφέρει μεγάλο μειονέκτημα. Ε, για παράδειγμα, εγώ ασχολήθηκα επανειλημμένα στο παρελθόν ε, με τον Frontex ε, και την έδρα της Βαρσοβίας και ο μισθολογικός λοιπόν συντελεστής και η μετατροπή που γίνεται στο πολωνικό ε, σημαίνει ότι τελικά οι εν λόγω εργαζόμενοι κερδίζουν πολύ λιγότερα χρήματα σε σύγκριση με τον προσωπικό των οργανισμών που έχει την έδρα τους σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λοιπόν τώρα λάβουμε υπόψη μας ε, και τον ε, προϋπολογισμό για τον οποίο, στον οποίο έχουμε προβλέψει και ε, μεγάλα πακέτα αμοιβών σε ό,τι αφορά τις, τα, τα, τα διευθυντικά επίπεδα του Frontex, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να διορθωθεί. Και κάτι ακόμα που αναφέρω στη γνωμοδίτηση μου είναι ότι τα κράτη-μέλη ε, φρόντιζαν στο παρελθόν να έχουν πάντοτε ένα εκπρόσωπο που θα συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια των λόγων αποκεντρωμένων οργανισμών. Ε, πράγμα βέβαια το οποίο είχε και κάποιες ε, φορές κομικά, κομικά αποτελέσματα όπου δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο είχε περισσότερα μέλη από ότι το σύνολο του προσωπικού του εν λόγου μικρού οργανισμού. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε ποια είναι η θέση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα του Συμβουλίου. Τα πράγματα βέβαια αλλάζουν όταν υπάρχει μια, ε, υπάρχει για παράδειγμα απόσπαση ενός ε, εργαζομένου από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή στι εργασίε τέτοιων οργανισμών, απέναντι στο οποίο είχε δείξει μια επιφυλακτική στάση το Συμβούλιο. Ε, θα μπορούσαμε λοιπόν ε, στο μέλλον να μπορέσουμε να προβούμε σε μια ερμηνεία, αν θέλετε και πάλι, των συνθήκων, ε, δηλαδή από την πλευρά των τριών θεσμικών οργάνων σε σχέση ε, με αυτούς τους αποτιτωμένους οργανισμούς. Μιλάμε δηλαδή εδώ για σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε μια, μια κοινή προσέγγιση, αφού δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστούν μέσα στις ίδιες τις συνθήκες. Και κάτι τέτοιο βέβαια συμπεριλαμβάνει ακριβώς και την απόσπαση από την πλευρά του Κοινοβουλίου ενός Ευρωβουλευτή που συμμετέχει ειδικότερα στα ε, διοικητικά συμβούλια ή στα διάφορα ε, συμβούλια ελέγχου των ελόγων οργανισμών. Αυτά από τη δική μου πλευρά και βέβαια είμαι ανοιχτό απέναντι στα σχόλια των ε, συναδέλφων. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για τι ε, επαγγελματικέ υπηρεσίε, ο οποίο μα ενημέρωσε όσον αφορά τα βασικά σημεία του σχέδιου γνωμοδότηση. Ποιο θέλει το λόγο, ο κ. Φερνάντε. Ευχαριστώ, πρόεδρε, να σα τα πω εκ μέρου του συναδέλφου Σαρβαμά που έχει αναλάβει το θέμα δεν μπόρεσε να παραστεί. Ζητεί να τον συγχωρήσετε. Ο κ. Σαρβάμα συμφωνεί με την γνωμοδότηση με το κείμενο Γκάιερ. Θέλω να σταθεί σε τρία σημεία. Πρώτα πρώτα όσον αφορά τον ε, συντελεστεί αυτό για τους μισθούς που θεωρείται θα πρέπει να διορθωθεί ούτω ώστε να αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος. Άλλο θέμα. Ο προπολογισμό των υπηρεσιών θα πρέπει να καταρτίζεται όπως προβλέπουν οι αρχές για την κατάρτιση προπολογισμού επί τη βάση τη απόδοση. Performance based budgeting. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τα έχουμε πει τόσε φορέ. Είναι η επανάσταση όσον αφορά την κατάσταση προπολογισμού. Δεν την είδαμε όμως ακόμα, ενώ αυτό υποτίθεται θα ήταν. Πάντω ελπίζουμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο παρά το ότι ο προπολογισμό τη Ένωση δεν είναι σαν τους εθνικούς προϋπολογισμούς και αυτό καμιά φορά το ξεχνούμε. Αφορά κάθε χρήση. Και δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι είναι 2% φέτος και στην επόμενη χρήση θα είναι 2% ε, του ΑΕΠ τέλο πάντων, του καθάριστου ε, χωρίου προϊόντος και την άλλη φορά μπορούμε κάτι άλλο. Τα ξέρουμε αυτά. Το τι προπηρεσμούς έχουμε όσον αφορά την αύξηση των ε, εισόδων. Καλά, τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι δικά μου. Είναι μια παρένθεση που την έβαλα στα, στα όσα ήθελε να δηλώσει ο κύριος Σαραβαμά. Τρίτον, όσον αφορά τα όσα θέλει να πει ο κύριος Σαραβαμά, είναι ότι πιστεύει πως θα πρέπει επίσης να ε, καταρτήσουμε, να αναδείξουμε τις προτεραιότητές μας για το έργο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Μια που θα πρέπει να αποφύγουμε επαναλήψεις, επικαλύψεις και έτσι να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη συνεργασία μεταξύ αυτών. Σας ευχαριστώ. Qui Άλλος θέλει το λόγο. Bien, monsieur Ευχόμαστε να είναι αυθεντικοί οργανισμοί αποκεντρωμένοι. Κύριε εισηγητά. Κάθε κράτος μέλος διεκδικεί ένα τέτοιο οργανισμό και ο καθένας προσπαθεί να τα τα ε, συμφέροντά του, τα εθνικά και που τέλος πάντων πάντοτε ε, έχω στο μυαλό μου το ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια αναδιάρθρωση, να έχουμε και έναν ευρωπαϊκό οργανισμό για την απασχόληση και για την επαγγελματική κατάρτιση και προσανατολισμό. Δύσκολο να φτιαχτεί ένας τέτοιος οργανισμός. Ε, κάποιοι οργανισμοί από αυτούς έχουν πλεονέκτημα όσον αφορά την πρικοδότηση, αλλά δεν μπορούμε όμως να περικόψουμε από την πρεκοδότηση των οργανισμών γιατί υπάρχει και το θέμα του ανταγωνισμού με τους εθνικούς αντίστοιχου οργανισμούς και οπότε γι' αυτό και λέω ότι συνήθως η κατανομή αυτών των οργανισμών δεν αφορά τόσο την ουσία αλλά εθνικούς εγωισμούς δεν είναι θέμα δηλαδή της ελεγγύης που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση κύριε Γκάιερ θέλετε να λάβετε το λόγο. Mm. 19 Δεκάτου στις 6 το απόγευμα θα καταδίνει οι τροπολογίες, 18 Δωδεκάτου θα ψήφουν στην Επιτροπή και στις 20 Δευτέρου του 19 θα ασχοληθεί η ΑΦΚΟ επί της ε, ουσίας για το κείμενό σας. Κύριος Γκάιερ. Με μεγάλη μου χαρά κύριε Πρόεδρε, η κατανομή λοιπόν των οργανισμών. Πάντοτε με διασκέδασε κάπως, ε, διότι είμαι και ιστορικός και ε, κάνω τη σύγκριση με πράγματα που συνέβαιναν τον Μεσαίωνα. λέω για να μην ε, ενοχλήσω κανέναν, η λέξη bastard, «bastardos» δεν είναι φρυσιά στα γερμανικά, τουλάχιστον όχι όπως στα αγγλικά. Όποιο λοιπόν θυμάται την ιστορία του Μεσαίωνος θα θυμάται τα μπάσταρδα παιδιά, δηλαδή τα νόθα παιδιά των δυναστιών που κάπως ενοχλούσαν. Το ίδιο με τους οργανισμούς. Όλοι χαίρονται που φτιάχνουν ένα καινούριο οργανισμό, όταν όμως πια αρχίσει να υπάρχει ο οργανισμός δεν τους ενδιαφέρει και τους ενοχλεί. Όταν πρόκειται να διδηθεί ένα οργανισμός, λοιπόν, σκοτώνονται οι χωρισμένοι, ποια θα πρωτοπάρει την έδρα. Εγώ χαίρομαι τώρα και εδώ και τι θα γίνει με την European Labour Authority. Θα γίνει μαχαίρωμα κανονικότατο για να αποκτήσουν την έδρα διάφορες χωρισμένοι. Και όταν θα ε, δουν ότι δεν έχουν κανένα οργανισμό, διότι υπάρχουν κάποιε χωρισμένοι που δεν έχουν κανένα οργανισμό, την έδρα του δηλαδή, στην επικράτειά του. Άλλε θα βγουν να πούν μα τι σημαντικό που είναι αυτό ο οργανισμό και οπωσδήποτε πρέπει να έχει την έδρα του δική του χώρα μέλη και δεν είναι καν θέμα χωρών μελών. Όταν ε, πρόκειται να μετακινηθεί η ΣΕΠΟΛ, η Ευρωπαϊκή Αστυνομία δηλαδή, η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε τότε να την στείλει σε ένα πραγματικά πολύ απομακρυσμένο τόπο. Θα ήταν λογικό ο οργανισμό αυτό να τοποθετηθεί στην Χάγη, διότι εκεί εδράζονται ήδη οργανισμοί με παρόμοια καθήκοντα. Τουλάχιστον θα είχαν υπάρξει έτσι κάποιες ε, συνέργειες. Α, ε, τώρα που έχει πάει στη Βουδαπέστη, είχε πάει σε πόλο και διάφοροι ευρωβουλευτές μάλιστα πάλεψαν ώστε ο οργανισμός πάντως να μην εγκατασταθεί στην Χάγη, να πάει στη χώρα τους, στη χώρα από την οποία προέρχονταν οι ίδιοι. Είναι ένα είδος δηλαδή του ενστήκτου του κυνηγού. Και βέβαια να μπορεί ο Ευρωβουλευτή να πει μετά, αν ναι, εγώ πάλεψα ώστε ο τάδε σημαντικό ευρωπαϊκό οργανισμό να έρθει στην πατρίδα μου, για παράδειγμα, στη δική μου έση. Και ανεξαρτήτως το αν είναι λογικό κάτι τέτοιο ή όχι. Έχω λοιπόν, εγώ πιστεύω, θεωρώ, ότι χρειάζονται όντω αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή τη έδρα ενό οργανισμού. Για παράδειγμα, η προσβασιμότητα. Πρέπει να πάρουν κοντά, α πούμε, μεγάλα αεροδρόμια. Ένα μεγάλο ε, διεθνή αερολιμένα. Για οργανισμού ιδίω που διατηρούν πολλέ επαφέ, όπω ο οργανισμό για τα φάρμακα ή τι χημικέ ουσίε. Πρέπει να πηγαίνουν πολύ εκεί για να κάνουν πιστοποιήσει των ουσιών αυτών. Άρα πρέπει ο οργανισμό αυτό να έχει την έδρα του κοντά σε ένα μεγάλο διεθνέ αεροδρόμιο. Ή να υπάρχει ένα διεθνέ σχολείο για τα τέκνα των υπαλλήλων που θα ε, τοποθετηθούν στον οργανισμό αυτό. Είναι δύο ας πούμε, βασικά αντικειμενικά κριτήρια τα οποία πρέπει να παίζουν ένα ρόλο στην επιλογή των εδρών. Αυτά σε ό,τι αφορά την κατανομή. Βλέπω τώρα ότι έχουμε τώρα και τους δύο οργανισμούς που έχουν την έδρα στο Λονδίνο μας των φαρμάκων υποτίθεται θα πάει να τοποθετηθεί στο Άμστερνταμ. Η Ολλανδική κυβέρνηση πάλεψε για να την αποκτήσει. Όταν όμως βγήκε η απόφαση για την αίμα, μπήκε όμως και το ερώτημα θα αναλάβει η Ολλανδική κυβέρνηση να πληρώνει και ένα μέρος των μισθωμάτων. Ξαφνικά έπιαψαν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ή πάντως χρειάστηκε να ασκηθεί πίεση ώστε να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους οι Ολλανδοί. Η δε Ιταλική κυβέρνηση δυσαρεστήθηκε με την επιχείρηση του Άμστερνταμ απέναντι στο Μιλάνο και συχνά μου λένε οι Ιταλοί συνάδελφοι τι ωραία που θα ήταν να οργανώσει αυτό δεν έχει τοποθέτηση στο Μιλάνο. Ποτέ δεν θα μπορέσει κανείς να τους ικανοποιήσει όλους, αλλά κάποια κριτήρια τέλο πάντων πρέπει να ισχύουν και να τηρούνται για τους ε, αποκεντρωμένους οργανισμούς. Για την κατανομή λοιπόν των οργανισμών ε, δεν μένουν πολλά πράγματα να πω ή να κάνουμε. Δεν νομίζω άλλωστε να χρειαζόμαστε και πολλούς άλλους οργανισμούς, εκτός πια και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλάβει ακόμα περισσότερα καθήκοντα, όπως τώρα με την οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων. Το ερώτημα είναι ποιο θα ελέγχει τα πράγματα αυτά. Εάν αποφασίσουμε εν τέλει ότι όντω θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, European Labour Authority, θα πρέπει να ενδυθεί το ένδυμα του οργανισμού και θα πρέπει να αποκτήσει κέντρα. Αυτό δεν θα σημάνει ωστόσο πληθωρισμό οργανισμών, κατά τη γνώμη μου. Μου φαίνεται ότι όμως έτσι απάντησα στις δύο ερωτήσεις σας. Α, ναι, μένει κάτι ακόμη. Εδώ οφείλω να επενέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πράγματι εξετάζει προσεκτικά εάν η νομική βάση στην οποία στηρίζεται ο οργανισμός όντως τηρείται για την ELA βλέπουμε για τον προϋπολογισμό ότι ορισμένα προγράμματα στο μέλλον θα εκτελούνται από την European Labour Authority, ELA. Θα αρχίσουν λοιπόν ήδη μεταφορές πιστώσεων στο πρόγραμμα, στον, ε, λειτουργικό προϋπολογισμό ή επιχειρησιακό προϋπολογισμό της ELA. Εγώ το βρίσκω σωστό αυτό και σας υποστηρίζω κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει δηλαδή η νομική βάση να είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένη υπάρχει και ένας οργανισμός που κινείται διεθνώς για την εκπαίδευση νεαρών ενηλίκων με έδρα στο Τωρίνο και κάποιοι που γνωρίζουν το θέμα αυτό και εθνικά. Νομίζω ότι και εκεί οι μέθοδοι είναι παρόμοιες. Θα μπορούσε και εκεί δηλαδή με κάποιο τρόπο να συγχωνευτεί. Αλλά για πάρτε την πρόταση που βάλετε την στην Επιτροπή Εξωτερικών θα σας πούν τότε ότι αυτό είναι ο μοναδικό μα οργανισμό και θέλουμε και εμείς να έχουμε έναν. Αν οι οργανισμοί είναι παιχνίδια των επιτροπών, έστω. Κάποια, κάθε επιτροπή έχει οργανισμούς με, τις, με τους οποίους συνεργάζεται πολύ στενά και σε βάση εμπιστοσύνη. Οι συνάδελφοι το θεωρούν, οι συνάδελφοι μας ευρωβουλευτές, θεωρούν ότι έτσι πάμε να τους πάρουμε κάτι να του αφαιρέσουμε κάτι όταν ερχόμαστε και ρωτούμε, μα είναι απαραίτητο ο οργανισμό, μήπω μπορεί η δουλειά να γίνει και διαφορετικά. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ κύριε Ισηγητά Άρα έχουμε το ραντεβού για τι ε, τροπολογίε. Κατάθεση το αργότερο στις 19 Νοεμβρίου στι 6 το απόγευμα. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στι 10 12 Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Χάουταλα η οποία όμως δυστυχώς δεν είναι παρούσα και εξέφρασε την επιθυμία να την εκπροσωπήσει ο κύριος Τάραντ για να εξηγήσει τα περί του σχεδίου γνωμοδοτήσεώς της, στο όνομα της δικής μας Επιτροπής, για συμφωνία αλίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Δημοκρατίας της ακτής του ελεφαντοστού. Κύριε Τάραντ, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος ε, καθώς ε, έχουμε ουσιαστικά μείνει τόσο λίγοι στην αίθουσα έτσι ώστε να είναι σαν ε, συνάντηση συντονιστών πλέον η συνεδρίαση μας. Ε, θυμάμαι πάντως η πρώτη έκθεση που είχα συντάξει για αυτήν την Επιτροπή αφορούσε μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ενεγάλης πριν από τέσσερα χρόνια και ουσιαστικά έκτοτε ε, το δικό μου όνομα ε, έχει γίνει αντικείμενο κατάρας ε, από την πλευρά τους αλλά και σε ό,τι αφορά τους Πορτογάλους, τους Ισπανούς και τους Σκοτσέζους ψαράδες. Σε κάθε περίπτωση η συνάδελφος μου ζήτησε να αναφέρω σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία μεταξύ δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ε, θα μπορούσε πραγματικά να μεταβάλει τι συνθήκε ζωή των αλλιών και των οικογενειών του. Ε, και γι' αυτό καλούμε την Επιτροπή να παραμείνει ε, σε επαφή με τι τοπικέ αρχέ, για να διασφαλίσουμε ότι κυρίω οι γυναίκε και εργαζόμενοι στον τομέα της επεξεργασία των ψαριών να είναι σε θέση να βελτιώσουν το εισόδημά τους και να συμβάλλουν ταυτόχρονα στην τοπική εκεί διατροφική ασφάλεια και την ανάπτυξη των κοινοτήτων αυτών. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε που μας τα διευκρινίσετε για το τι θέλει να προτείνει η κυρία Χάουταλα με το σχέδιο γνωμοδότησης. Οι συνάδελφοι που άντεξαν μέχρι τώρα θέλουν να πούν τίποτα. Όχι κύριε Γκρατιδάπα, λέω ότι είναι τέλεια η έκθεση. Δεν επιδέχεται παρατηρησία, ε, άρα θα πρέπει να διαβιβάσετε αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκρατιδάπα στην κυρία Χαουταλά. Έτσι όπως μας τα είπε ο κύριος Ταράντ, πάντως ε, ήταν ε, πάρα πολύ πιστικά. Αν κανείς δεν θέλει το λόγο, τότε θα σας πω το μυστικό για τις τροπολογίες. 9 11 το μεσημέρι, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή. Και η ψήφιση θα γίνει στις 10-12 αλλά στην Επιτροπή, αλλιές που είναι κυρίως αρμόδια Επιτροπή, θα γίνει στις 23 πρώτου. Θα πάει δε το θέμα στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Άρα πριν τις εκλογές θα έχουμε την κύρωση της εν λόγω ε, εμπορικής αλληλευτικής συμφωνίας. Τελειώσαμε τα θέματα της σημερινής διάταξης, συνάδελφοι. Θέλω να σας πω επίσης ότι θα τα ξαναπούμε 21 και 22 Νοεμβρίου, οπότε και θα ψηφίσουμε τι, τι είπατε, κάτι λέει στον πρόεδρο η, η γραμματέας. θα ψηφίσουμε τις γνωμετίες που συζητήσαμε σήμερα, οπότε και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εξέταση των γνωμετήσεων που εκκρεμούν. Και άρα όλα αυτά θα γίνουν 21 και 22 Νοεμβρίου. Στις 27 Νοεμβρίου έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και θα επανέλθουμε στα θέματα κράτους δικαίου, Στην αναγκή προστασία του στη Αξίας της Ένωσης, στις 3 Δωδεκάτου δε, έχουμε το Invest EU, στην κοινή συνεδρίαση με την Οικονομική Επιτροπή που θα έχουμε και θα έχουμε επίσης και τα θέματα τα σχετικά με την θωράκιση της Ευρωζώνης. Στις 10 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο πρόκειται να έχουμε μία συνεδρίαση έκτακτη επιπλέον και θα είναι η τελευταία για το 18 πάρα πολύ σπουδαία στιγμή επομένω. και τώρα συντονιστές και σκιώδεις ε, εισηγητέ θα πρέπει να έρθουν εδώ στις 6 για να γίνει η πρώτη συνάντηση ε, προπαρασκευαστικού χαρακτήρα και τη συνδιαλλαγή όσον αφορά το σχέδιο του 19. Η ιδέα η υπεύθυνη κομματική πειθαρχία αλλά και η βοηθή, θα πρέπει να το θυμίσουν σε αυτούς που οφείλουν να ε, είναι εδώ που θα πρέπει να πάνε και στην Επιτροπή της Συνδιαλλαγής που είναι ο ρόλος τους ακριβώς η τακτή παρακολούθηση, η παρουσία για να υπάρχει την κρίσιμη στιγμή απαρτία. Donc nous nous retrouvons dans cette salle à 17h45 pour 6 παρατέταρτο για την προπαρασκευαστική συνάντηση. Et ayant lieu après-demain matin à 9h. 9 η ώρα θα γίνει η πρώτη συνάντηση συνδιαλλαγής. Αύριο.